ότι προέκυψε κάτι από αυτή την έκθεση το οποίο θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Δεν θα τελειώσουμε με την ψηφοφορία. Ευχαριστώ.